Συνάδελφοι, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Παίζαμε μουσικές καρέκλες στην Επιτροπή. Έπρεπε να μετακινηθούμε το απόγευμα. Οπότε πάμε κατευθείαν στην ε, υιοθέτηση της σημερινής διάταξης. Έχω μία τροποποίηση να προτείνω. Το σημείο για αύριο, για τους Γεζίντι, έχουμε κάποια νέα, δεν έχω και τις σημειώσεις μου, είναι το σημείο 14 για τους γεζίδες στο Ιράκ. Αναβάλλεται η κατάσταση των γεζίδες στο Ιράκ. Αύριο το απόγευμα θα το συζητούσαμε. Θα αναβληθεί γιατί ο βασικός ε, εισηγητής δεν έχει πάρει βίζα. Δεν έχει θεώρηση ακόμη, οπότε θα μπορέσουμε να κάνουμε τη συνάντηση αυτή κάποια στιγμή άλλη. Άρα θα τελειώσει πιο νωρί η συνεδρίασή μα αύριο το απόγευμα. Σημειώστε λοιπόν παρακαλώ ότι κάνουμε αυτή την αλλαγή στην ημερησία διάταξη για αύριο. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, κάποιε ανακοινώσει. Η 8, η 8 Μαρτίου καταρχάς είναι η Διεθνής ημέρα της γυναίκας και το φέτος η εκστρατεία ονομάζεται Balance for Better. Αύριο το πρωί θα κάνουμε μια συζήτηση για το σχέδιο δράσης που θέλει να προωθήσει αυτή την ε, ισορροπία για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Ελπίζω να είσαστε παρόντες στην ανταλλαγή αυτή απόψεων για να μπορέσουμε να εορτάσουμε την 8η Μαρτίου, την Διεθνή ημέρα της γυναίκας. Δεύτερο σημείο, δυστυχώς πρέπει να μιλήσουμε για τον Brexit, δυστυχώς για μένα. Με ρωτούν οι συνάδελφοι τι γίνεται. Ε, ακόμη δεν ξέρουμε τι γίνεται. Υπάρχει ε, αβεβαιότητα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η βασική ψηφοφορία θα γίνει 12 και 13 Μαρτίου τώρα. Ε, και εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω ότι είμαστε εδώ ένα μήνα πριν την 21 η Μαρτίου και δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει, για μας αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι ότι όντως, παρόλο που έχουμε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο πολύ μεγάλη ασάφεια και βεβαιότητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκινά τη δική του διαδικασία, δηλαδή την παροχή συγκατάθεσης για την Συμφωνία Αποχώρησης. Η Επιτροπή Στεγματικών Υποθέσεων, η ΑΦΚΟ, προετοιμάζει μια σύσταση ε, που θα αποτελέσει την βάση για την δική μας συγκατάθεση. Ε, υπάρχουν διάφορα ψηφίσματα, ε, όπως και αυτά, και αυτή η γνωμοδότηση θα, έχει, θα είναι ναι ή όχι. Μπορεί να αλλάξει βέβαια η απόφαση, αλλά προς το παρόν θα δοθεί είτε θετική είτε αρνητική απάντηση. Κάποιες επιτροπές που έχουν να θίξουν διάφορα θέματα, θα στείλουν στην ΑΦΚΟ τις θέσεις τους, το ζήτησε η ΑΦΚΟ για τον Brexit, για να μπορέσουν από τους, από πρόεδρους των ε, επιτροπών αυτών να πάνε στον πρόεδρο της ΑΦΚΟ, αλλά προς το παρόν δεν έχει αποσταλεί κάτι. Το ψήφισμα αυτό θα έχει να κάνει μόνο με την ε, συμφωνία αποχώρησης, όχι για τις μελλοντικέ σχέσεις με το Ηνωμένο και η διαδικασία δεν μας επιτρέπει να θέσουμε κάποιο θέμα ε, ε, οπότε εμείς δεν θα στείλουμε τέτοια επιστολή στην Επιτροπή ΑΦΚΟ. Αν αυτό βεβαίω αλλάξει, η Επιτροπή θα μπορέσει να θέσει τα οποιαδήποτε ζητήματα στην γενική συζήτηση που θα γίνει τότε. Αυτά έτσι ενημερωτικά για το τι γίνεται με τα τυπικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρμογή του Brexit και της Συμφωνίας Αποχώρησης. Εντάξει, Ωραία. Ε, σημείο 4. Έγκριση των ε, πρακτικών. Έχουμε πρακτικά 8η-9η ε, Οκτωβρίου, 12η Νοεμβρίου, 19η 20 Νοεμβρίου, 13η Δεκεμβρίου. Αν έχετε σχόλια, παρακαλώ μέχρι το τέλο τη συνεδρία τα σχόλιά σα στη γραμματεία, γιατί αλλιώ θα θεωρηθούν ω ε, εγκεκριμένα. Σημείο 5. Ανακοινώσει από την Κομισιόν. Έχει η Κομισιόν να μα ανακοινώσει κάτι. Παρακαλώ, σα ακούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα κάτι ενημερωτικό. Θα το ξέρετε, αλλά να σας επιστήσω προσοχή στο εξή. Οι Ευρωπαϊκές ημέρες ανάπτυξης 18 και 19 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του Τούρε Ταξί. Ε, βασικό θέμα είναι οι ανισότητες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως πάντα προσκαλείται να οργανώσει μια σύνοδο και βεβαίως Όλοι είσαστε καλοδεχούμενοι, είστε ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε στις ε, δραστηριότητες. Για να σας δώσω μια μικρή γεύση για το τι έγινε πέρσι. Είχαμε περίπου 8.000 ε, συμμετέχοντες και 1.200 ε, οργανισμούς που συμμετείχαν. Είναι πραγματικά σημαντικό το, σημαντική εκδήλωση αυτή για την ανάπτυξη. Και βεβαίω οι επίσημε πληροφορίε, οι προσκλήσει κτλ. θα ακολουθήσουν. Απλώ ήθελα να σα το υπενθυμίσω. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Από την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ κάτι. Όχι. Εντάξει. Ωραία. 18-19 Ιουνίου, μετά τις ευρωεκλογέ δηλαδή, οπότε φαντάζομαι ότι περισσότεροι ευρωβουλευτές ε, θα είναι μέλη της ε, των Επιτροπών, γιατί θα είναι μέλη μέχρι την 1η Ιουλίου, οπότε φαντάζομαι ότι θα μπορούν οι τρέχοντες ε, βουλευτές να συμμετάσχουν, γιατί ε, για να οργανώσουμε κάτι θα είναι μάλλον δύσκολο, αλλά για να συμμετάσχουμε ε, είναι λίγο πιο απλό. Όντω, όπω είπατε, είναι σημαντικέ οι μέρε αυτέ ανάπτυξη. Δυστυχώ φέτο είναι λίγο το χρονοδιάγραμμα πιεσμένο. Λοιπόν, πάμε στο σημείο 6, που είναι σημαντικό για τα συνοδευτικά μέτρα για την μπανάνα. Θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων με, τον, με την αυτού εξοχότητα, τον κύριο Ντανιέλ Εβίνα Αμπέ, που είναι ο πρέσβης του Καμερούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, ο πρόεδρος της ε, ομάδας εργασίας για την μπανάνα από τις χώρες ΑΚΕ. Ε, καλώς ήρθατε, κύριε πρέσβη. Ε, αυτές τις, ε, αυτό το θέμα το έχουμε συζητήσει εμείς, το θέμα της μπανάνας και των μέτρων για όσους πήγατε στην Σύνοδο στην Αμπιτζάν, ε, επίσης έγινε μια πολύ καλή αποστολή, μια επίσκεψη για να δούμε μπανανοφυτίες και παραγωγή μπανάνα στην Αμπιτζάν και ξέρουμε πραγματικά πόσο σημαντική είναι η βιομηχανία μπανάνας σε πολλές, ε, για πολλές χώρες ΑΚΕ. 1,4 τόνοι μπανάνας ε, παράγονται κάθε χρόνο και ένα μεγάλο κομμάτι των, εξο, των έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ένα ειδικό πρόγραμμα συνοδευτικών μέτρων για την μπανάνα για να βοηθήσει τις ε, εταιρείε και τις χώρες που ε, εμπορεύονται μπανάνα ε, μετά τις αλλαγές που έγιναν στην αγορά μπανάνας λόγω των, της απόφασης του ΠΟΕ ότι η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να αλλάξει τους δασμούς για τις μπανάνες. Οπότε τα συνοπτικά αυτά μέτρα ήταν ε, κομμάτι της ε, συμφωνίας της Γενέβης για την, εμπορία, για την εμπορία των μπανανών και επιτέλους λύθηκαν διάφορες διαφορές που υπήρχαν εδώ και 15 χρόνια με αυτή την απόφαση. Αυτό που θέλουμε τώρα να μας πει ο κύριος Πρέσβης είναι πώς ή αν βοήθησαν τα μέτρα αυτά στα συνοδευτικά, τις μπανάνες, για τις, ε, τις χώρες ΑΚΕ να προσαρμοστούν σε αυτό το νέο καθεστώς δασμών. Και αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρξει στήριξη στις μπανάνες και στις χώρες παραγωγής τους. Βεβαίως έχουμε ένα νέο χρονοδιάγραμμα για την ε, συνεργασία και την ανάπτυξη για το 2021. Η Κομισιόν συζητά, θα συζητήσει μάλλον ε, το θέμα αυτό τις επόμενες εβδομάδες, οπότε ε, μπορούμε τώρα να ενημερωθούμε, να δούμε πού βρίσκεται η κατάσταση με το BAM, τα μέτρα δηλαδή τα συνοδευτικά, και τι γίνεται με τις χώρες, ας πούμε, όπως ε, το Καμερούν, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Γκάνα, η, η Τζαμάικα, η Αγία Λουκία, η Γραναδίνη, το Σουρινάμ, μεγάλες χώρες παραγωγών ε, μπανάνας. Εγώ έχω δει στο ε, πράσινο κροτήρι ε, παραγωγή μπανάνας, στον Άγιο Βικέντιο πολλά χρόνια πριν και ξέρω ότι πραγματικά είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας αυτός για πολλούς ε, γεωργούς και για πολλές χώρες. Οπότε κύριε Πρέσβη, με χαρά θα ακούσουμε όσα έχετε να μας πείτε. Merci, euh, Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε ευτυχείς που διαπιστώνουμε ότι σε διάρκεια ε, τριών μηνών η ομάδα ΑΚΕ στις 30 Ιανουαρίου ήταν εδώ στην Επιτροπή σας για τη ζάχαρη και σήμερα για την μπανάνα για δεύτερη φορά. Όπως είπατε είμαι ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας για την μπανάνα και θα προσπαθήσω να παρουσιάσω κάπως κάποια στοιχεία που ε, θα μας επιτρέψουν να συζητήσουμε ε, ε, με στοιχεία. Ο τομέα τη Μπανάνα, κυρία Πρόεδρε, εξακολουθεί να αποτελεί έναν παράγοντα ε, πλούτου ε, για τις χώρε ΑΚΕ. 30.000 θέσεις άμεση εργασία και 50.000 έμεσε. είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί αυτός ο τομέας λόγω και του πολλαπλασιαστικού του ΕΦΕ. Το είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οθέτησε συνοδευτικά μέτρα για την ε, μπανάνα, τα BAM, η ΜΑΜΠΑ, ανάλογα με την γλώσσα, είναι, ε, αφορούν πολλές χώρες και φτιάχτηκαν για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να ενθαρρυνθεί η ε, διαφοροποίηση. Η ομάδα και ε, παραμένει όμως ανήσυχη όσον αφορά την αντιγωνιστικότητα του τομέα της μπανάνας στην ευρωπαϊκή αγορά δεδομένη της ε, ε, του γρήγορου ρυθμού των περιφερειών προτίμησης που έχουν ξεπεράσει τα μέτρα προστασία, τα συνοδευτικά μέτρα τα οποία ε, ανέργονταν σε 190 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από τη Συμφωνία της Γενέβης ε, του ΠΟΕ του 2009, η Συμφωνία Σύνδεσης ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής και η παραγωγή της Λατινικής Αμερικής έχουν φτάσει σε συσσωρευμένες οικονομίες της τάξης του 1,9 δις ευρώ όσον αφορά δασμούς. Αυτό ε, αφορά την παραγωγή της Λατινικής Αμερικής και κατά συνέπεια υπήρξε μείωση δραστική της ε, τιμής της ε, χονδρικής μέχρι και 20%. Πράγμα το οποίο επιβαρύνει τις χώρες ΑΚΕ, των οποίων το περιθώριο είναι πολύ ευαίσθητο σε τέτοιου είδους διακυμάνσεις, τόσο μεγάλες διακυμάνσεις. Αυτά καλύφθηκαν εν μέρη από τα συνοδευτικά μέτρα. Οι χώρες της Κεντρικής και ε, Λατινικής Αμερικής ε, επικρατούν στην αγορά γιατί έχουν αυξήσει το συνολικό τους μερίδιο του 69,9% της ε, αγοράς το 2016 έχουν φτάσει στο 75% ε, φέτος, δηλαδή τεράστια αύξηση εντός δύο ετών, ενώ η παραγωγή τους έχει πέσει κατά 3 περίπου της 100. Πρόσφατα, οι εισαγωγέ από την Ικαράγουα, το Περού και την ε, Γουατεμάλα ε, γνώρισαν ακόμα μια σημαντική αύξηση και έχουν ξεπεράσει τα κατόφλια που έχουν θεσπιστεί για τις χώρες αυτές μέσα στο πλαίσιο του μηχανισμού σταθεροποίησης, πράγμα το οποίο είχε αρνητικές επιπτώσεις στην τιμή της αγοράς. Η παραγωγή και Ανησυχούν λοιπόν λόγω αυτής της μεγάλης αύξησης εισαγωγών από τις χώρες της ε, Λατινικής Αμερικής. Έχουμε σε σημείο ε, ε, εξόδου της ε, μπανάνας των χωρών ΑΚΕ από την ευρωπαϊκή αγορά. Ωστόσο, ο μηχανισμός δεν μπόρεσε να, να αντιδράσει όσον αφορά τις υπερβολικές ε, ε, εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε πως ε, θα εφαρμοστούν οι κανόνες με μεγαλύτερη αυστηρότητα όσον αφορά την υπέρβαση των κατοφλίων και τις συνέπειές τους που θα παραταθούν πέρα από το 2019. Κυρία Πρόεδρε, το σενάριο το οποίο σας περιέγραψα αποτελεί άμεση απειλή και ζωτική σημασία απειλή για τον τομέα της μπανάνας των χωρών και είναι απαραίτητο να φτιαχτεί ένας επιπλέον μηχανισμός στήριξης πέρα από το 2019. Με ρωτήσατε ήδη αν θα πρέπει να συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης στην μπανάνα. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τη στήριξη στον τομέα της μπανάνας ώστε να καταστεί πιο ανταγωνιστικό στις διεθνείς αγορές διατηρώντας ε, και αυτό το μοντέλο. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η στήριξη προς την μπανάνα ήταν αποτελεσματική στο βαθμό που αυτή η στήριξη επέτρεψε καλά αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, την ανάπτυξη ε, αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διαφοροποίηση, την μεταποίηση, την παραγωγικότητα και την υλοποίηση και αύξηση των εσωτερικών αγορών. Ωστόσο, θα πρέπει να μεριωθούν ακόμα τα κόστη και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα μέσω κατάλληλων μέτρων καταπολέμηση των νόσων, πρόσβαση στι πιστώσει για του γεωργού, μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στι περιοχές τη υπαίθρου που είναι οι πιο ευάλωτε. Με ικανοποίηση, ωστόσο, διαπιστώνουμε την επιστολή με ημερομηνία 20 Μαρτίου 2018 που μετέφερε ο Επίτροπος Εμπορίου όπου ε, καλεί για τη συνέχιση των ε, ισχυών των προσπαθειών μέσω της ε, ρύθμισης συνεργασίας όπου στηρίζεται και ο ιδιωτικός τομέας με τα... μέσα στο οποίο είναι και τα μέτρα για τη στήριξη της μπανάνας. Κυρία Πρόεδρε, οι παραγωγή μπανάνας της Αφρικής έχουν δώσει συνέχεια στην έκκληση αυτή της Επιτρόπου Εμπορίου και ξεκίνησαν ε, διαπραγματεύσεις με τα μέλη τους και έχουν επεξεργαστεί μια στατικική ανάπτυξη για τον τομέα. Έχουν καλέσει μάλιστα τους ομολόγους τους της περιοχής της Καραβικής να κάνουν το, το ίδιο, λαμβάνονταν υπόψη τι ιδιαιτερότητές του. Αυτή η πρωτοβουλία οδήγησε στην εκπόνηση ενός λευκού βιβλίου για την Αφρικανική μπανάνα που στόχο έχει να παρέχει ουδέτερα, ουδέτερη βάση δεδομένων ώστε να μπορέσουν να τη μελετήσουν οι θύνοντες και οι αρμόδιοι για την λήψη αποφάσεων. Στόχο έχουν όχι μόνο τη αντιμετώπιση του ανταγωνισμού από τους λατινοαμερικανούς ε, ε, παραγωγούς, αλλά ώστε να θεσπίσει μια βάση ε, ανταγωνιστικό, ανταγωνιστική υπέρ των Αφρικανών παραγωγών. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να σας δώσουμε, αν χρειάζεστε, επιπλέον πληροφορίες για τις λύσεις που προτείνονται μέσω αυτού του στρατηγικού σχεδίου. Εξάλλου, Ενημερωθήκαμε με ανησυχία ότι στη διάρκεια της πέμπτης ετήσιας συνεδρίασης της Κομισιόν για το εμπόριο και τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η σημερινού Περού που έγινε στο Κίτο αυτές οι τρεις χώρες ζήτησαν ε, πλήρη απελευθέρωση του τομέα της μπανάνα που ξεκίνησε ε, το 2009 και ζητούν να είναι ε, αδιαφοροποιητές οι διασμολογικές συνθήκες για την μπανάνα των χωρών ΑΚΕ. Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε μαζί σας για να βρούμε λύσεις και να αντιμετωπίσουμε τα κολοσσία προβλήματα που αντιμετωπίζει η μπανάνα των χωρών ΑΚΕ σε εμπορικό επίπεδο, αλλά για να μπορέσουμε και βιώσιμα να συμβάλλουμε στις διάφορες χώρες. Ζητούμε λοιπόν το πρόγραμμα για τα συνοδευτικά μέτρα της μπανάνας να συνεχιστεί και να ενισχυθεί. Επιπλέον καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Επιτροπής σας να διατηρήσει την υπόσχεση που ανέλαβε, ε, δηλαδή τη διατήρηση μιας σταθερής τιμής των 75 ευρώ τον τόνο. Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συνεργασία θα μπορέσουμε να βρούμε ε, ε, θετικά εμπορικά μοντέλα ώστε να μην βαθύνει η ρήξη και να ευνοήσουμε έτσι έναν ισότιμο κόσμο. Πριν να, να σταματήσω θα σας πω το εξής και θα διευκρινίσω το εξής. Όταν λήφθηκαν τα μέτρα το 2009, οι χώρες ΑΚΕ συνέχισαν να χαίρουν μέτρων για την μπανάνα τρία χρόνια αργότερα. Και αυτά τα τρία χρόνια ποτέ δεν καλύφθηκαν. Δηλαδή, λειτουργήσαμε σαν αυτά τα τρία χρόνια να είχαμε συνοδευτικά μέτρα, ενώ αυτό δεν ίσχυε. Μέσω της ομάδας εργασίας προσπαθήσαμε να τα παρατείνουμε, αλλά δεδομένων των προβλημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορέσαμε. Ήθελα λοιπόν αυτό να το τονίσω, διότι έτσι Κάποιοι μπορεί να βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο, αλλά πιστεύω πως είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει κανείς να έχει υπόψη του πριν να προβεί σε αξιολόγηση των έσων έχουν γίνει. Σας ευχαριστώ. Ε, με συνοδεύει ένας εκπρόσωπος των παραγωγών και έπειτα από τη γραμματεία της ΑΚΕ με τους οποίους παρακολουθούμε το θέμα αυτό στο επίπεδο της γραμματείας της ΑΚΕ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όταν συναντηθήκαμε στο Αμπιτζάν είχαν οργανώσει αυτές οι εταιρείε παραγωγής μπανάνας ε, ε, μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Όταν βλέπει κάτι κανείς με τα δικά του μάτια δεν το ξεχνάει εύκολα. Είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό. Τώρα θα ακολουθήσουμε μια κάπω ε, διαφορετική διαδικασία. Πριν δώσω το λόγο στα κράτη-μέλη, θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι ακούσαμε κάποια πράγματα από τον πρέσβη. Ε, ακούσαμε ότι η αύξηση των εισαγωγών από τη Λατινική Αμερική που, που, έχει να κάνει με τις εμπορικές συμφωνίες όπως αυτές με το Περού φαντάζομαι. Αυτό έχει επιπτώσει λοιπόν στις τιμές. Ε, γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε κάτι δηλώσεις ε, πέρυσι για το, τις κοινέ ε, κοινού ελληνικού δασμού για τι μπανάνε. Ε, Μόλι επέτρεψα από τη Σενεγάλη. Ε, είναι γνωστή η επιθυμία μα ε, να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τις θέσει εργασία στην Αφρική. Ε, καλό θα είναι λοιπόν η Κομισιόν να μα πει πού βρισκόμαστε στο συνεφορά το θέμα αυτό. Ποια σχέδια έχουμε. είτε με τον Τίκη είτε με άλλα όργανα. Είναι ο κ. Ντεκνόπ εδώ νομίζω είναι και η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου όμως αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω ποιος θέλει το λόγο πρώτος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μας δίνετε το λόγο, το λόγο πρώτους. Εμείς προφανώς και θα ακούσουμε τις απόψεις όλων, βεβαίως, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Θα απαντήσω σαφώς στα δύο κεντρικά ερωτήματα μετά την παρουσίαση του κυρίου Πρέσβη, μια παρουσίαση η οποία αποτυπώνει ε, σαφώς και τις δικές μας ανησυχίες, ε, τις κοινέ μας ανησυχίες, όταν ακούμε δηλαδή για υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας ε, αλλά και τη διαφοροποίηση στον κλάδο αυτό στις χώρες ΑΚΕ ε, και ότι για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει βεβαίως να λάβουμε υπόψη μας ε, και τον ιδιωτικό τομέα και να δώσουμε έμφαση και στην κλιματική αλλαγή. Εμείς δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με όλες αυτές τις ανησυχίες. Τώρα στην πράξη, σε ό,τι αφορά την διεθνή συνεργασία και τις σχετικές συμφωνίες με τις χώρες αυτές, αυτό σημαίνει το εξή. Όταν δεν είναι στην ημερήσια διάταξη να εργαζόμαστε ε, για, και να μιλάμε για τη δεύτερη φάση του προγράμματος BAM, ε, ακούσαμε τον πρέσβη που είπε ότι είτε θα έχουμε μια δεύτερη φάση είτε θα πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι υποστήριξης. Αυτό είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε και εμείς. Λέμε λοιπόν σαφέστατα ότι είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συνέχιση της υποστήριξης των χωρών που το επιθυμούν και στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν διάφορες διαδικασίες που μας επιτρέπουν να θεσπίσουμε προγράμματα υποστήριξης του κλάδου και άλλων κλάδων, εφόσον το επιθυμούν, το επιθυμούν κάποιες χώρες, κάποιες εθνικές αρχές. Ε, και είμαστε κοντά στο τέλος ενός κύκλου, πρέπει να ετοιμάσουμε τον επόμενο, οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτή Αυτό είναι που μπορούμε να πούμε σήμερα, δηλαδή να συμβουλέψουμε τις εθνικές αρχές των χωρών αυτών να έρθουν σε επαφή με τους εκπροσώπους μας εκεί, επιτόπου, έτσι ώστε να έχουμε αυτήν την κοινή προσέγγιση, το κοινό όραμα για την υποστήριξη του κλάδου. Αυτά για το, κλάδο, το, το, σκέλος που αφορά τη συνεργασία. Και το δεύτερο ερώτημα που θέσατε, Πρόεδρε, ε, πολύ σωστά θυμήσατε την επιστολή της 28ης Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, του 2018, της Επιτρόπου Εμπορίου. Ε, το περιεχόμενο της επιστολής αυτής βεβαίως είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή που ε, να ε, μας κάνει να μπορούμε να πούμε λοιπόν, ή να σκεφτούμε ότι αυτά που αναφέρουν στην επιστολή αυτή δεν θα γίνουν σεβαστά. Αυτή είναι η γραμμή μας ε, και σε επίπεδο εμπορικής πολιτικής και σε επίπεδο βοήθειας για την ανάπτυξη, αναπτυξιακής βοήθειας. Ε, αυτά θέλω να πω, έτσι και να κλείσω θετικά και αναμένουμε να ακούσουμε τις απόψεις των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ήταν όντω χρήσιμο να ακούσουμε αυτή την επιβεβαίωση ότι δεν έχει αλλάξει η πολιτική. Λοιπόν, ποιο θέλει το λόγο, Γενική Διεύθυνση Trade ίσω ή σα κάλυψε. ή σας κάλυψε, η ντευκο σα κάλυψε, πολύ ωραία. Ποιο θέλει το λόγο, και εγώ έχω ένα ερώτημα, αλλά πρώτα ο Νόρμπερτ. <clears throat> Ε, Ευχαριστώ. Περισσότερα ερωτήματα έχω αντί για απαντήσεις, γιατί το θέμα αυτό μου φαίνεται να είναι πολύ περίπλοκο. Θα προσπαθήσω να κάνω μια περίληψη καταρχάς, έτσι όπως τα κατάλαβα αυτά που ακούσαμε. Υπάρχει στήριξη ακόμη για τις χώρες ΑΚΕ που παράγουν μπανάνες και αυτή η στήριξη κάποια στιγμή θα εκπνεύσει. Θα υπάρξει δηλαδή μια φάση 2 όπως ακούσαμε ή τέλο πάντων θα υπάρξουν και άλλες συμφωνίες έτσι ώστε οι χώρες που έχουν πολλές εξαγωγές μπανάνας να μπορούν να στηριχθούν. Καλό είναι που οι χώρα ΣΑΚΕ είναι μαζί και εμείς εδώ σε Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να κάνουμε συμφωνίες με τις χώρες ΑΚΕ για το πώς μπορούμε στο μέλλον να ορίσουμε τον, και να στηρίξουμε τον τομέα της μπανάνας στο μέλλον μέσω των ε, συνοδευτικών μέτρων. Κύριε Πρέσβη, μιλήσατε για τη στήριξη 75 ε, ευρώ τον τόνο της μπανάνας. Αυτό είναι το ποσό που πληρώνετε τώρα και θεωρείτε ότι η στήριξη και στο μέλλον θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο, ανεξάρτητα από τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει αυτή η στήριξη. Δεύτερο ερώτημα. Οι χώρες ΑΚΕ βρίσκονται σε ανταγωνισμό με τους χώρες εξαγωγούς ε, εξω, εκτός χωρών ΑΚΕ, δηλαδή η Λατινική Αμερική και η Κεντρική Αμερική. Και σημειώσατε ότι εκεί η ισορροπία είναι κάπως αρνητική για τις χώρες ε, ΑΚΕ. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι μπορεί να γίνει ώστε να ξαναυπάρξει ισορροπία, ώστε οι χώρες ΑΚΕ που είναι οι πιο φτωχές χώρες κατά κανόνα σε σχέση με την Κεντρική Αμερική και την Νότιο Αμερική τι μπορεί να γίνει λοιπόν από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε αυτές τις χώρες, ΑΚΕ, να μπορέσουμε να τις στηρίξουμε επικοδομητικά. Ευχαριστώ, Νόρμπερτ. Ένα ερώτημα και από μένα, κύριε Πρέσβη. Στην εισαγωγική μου παρέμβαση μίλησα για το Brexit και τα όσα συμβαίνουν, αλλά το Brexit θα επηρεάσει και την βιομηχανία μπανάνας από τις χώρες ΑΚΕ. Έλεγξα κάποια αριθμητικά στοιχεία. Είπατε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι περίπου το 20% των συνολικών εισαγωγών Ευρώπη, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα τρίτο των μπανανών έρχονται από χώρες ΑΚΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, η ομάδα σας έχει συζητήσει το θέμα του Brexit και ποιο αντίκτυπο θα έχει και αν θεωρείτε ότι μπορούν να υπάρξουν κάποια ευρωπαϊκά μέτρα ειδικά για την κατάσταση του Brexit. Βεβαίως, ακόμη στη φάση αυτή δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος που θα ξεκινάει από τον Απρίλιο ή 30 Μαρτίου, με πάση περιπτώσει, οπότε θα υπάρξει περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστεί κανεί για τι διάφορε αλλαγέ. Εγώ ελπίζω ότι θα υπάρξει μεταβατική περίοδο. Τουλάχιστον η μεταβατική περίοδο, αν όχι τίποτε άλλο. Αλλά θα με ενδιαφέρε να ακούσω τι πιστεύετε για τον Brexit και πώ μπορεί να επηρεάσει την μπανάνα. Ε, νομίζω ότι δεν έχω η Κομισιόν άλλα ερωτήματα, οπότε σας ακούμε. Και βεβαίω μπορείτε να απαντήσετε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ξεκινήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή βέβαια δεν έθεσε ερωτήματα. Σε μεγάλο βαθμό επιβεβαίωσε αυτά που είπα ε, και νομίζω ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες μας. Στη δήλωσή μου άλλωστε αναφέρθηκα στην επιστολή της Επιτρόπου. Ήμουν σαφής δεν θέλουμε φάση 2 σε ό,τι αφορά τις ε, πληρωμές. Εμείς ε, εδώ θεωρούμε, συμφωνούμε μάλλον να ε, συμμετάσχει και ο ιδιωτικός τομέας στο θέμα αυτό της μπανάνας, εμείς ως χώρες ΑΚΕ. Αυτό όμως που θέλουμε είναι να, συνεχίσει, να συνεχιστεί η στήριξη της μπανάνας. Δεν θέλουμε να βγει δηλαδή εκτός ατζέντα ο φάκελος αυτός. Ο Υπουργός Εμπορίου μας είπε ότι αν συμβεί αυτό ουσιαστικά είναι σαν να εργανώνουμε μια πρώτη τάξη ως κηδεία στην μπανάνα το χρόνο και. Λοιπόν, και τα 75 ευρώ τον τόνο. Αυτό είναι μια εξέλιξη. Ε, το έχουμε πει και στο παρελθόν και η Κομισιόν, ε, σύμφωνα με τους παραγωγούς μας, Εάν το κατόφλι των 75 ευρώ ανατόνο κατέβει πιο κάτω, μιλάμε για το τέλος του τομέα αυτού της μπανάνας στις χώρες ΑΚΕ. Είχε αναλάβει αυτή την δέσμευση η Κομισιόν. Ελπίζουμε λοιπόν και επιθυμούμε αυτή η απόφαση να παραμείνει. αυτό το 75 ευρώ είναι ένα κατόφλι. Αν πάμε κάτω από το 75, τελείωσε. Δεν μπορούμε πια να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και τα συνοδευτικά μέτρα στην μπανάνα, όπως τα ζητάμε εμείς, Γι' αυτό και στην αρχή είπα ότι εμείς δεν επωφεληθήκαμε αυτών των μέτρων για τρία χρόνια. Τρία χρόνια καθυστέρηση δηλαδή έχουμε. Βεβαίω, δεν έχω κάποια μαγική σφαίρα, αλλά αν εντό των τριών αυτών ετών είχαμε αυτά τα μέτρα, μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είμαστε σίγουροι, αλλά μπορεί να ήταν διαφορετικά. Ήθελα λοιπόν να το πω αυτό για να εξηγήσω την υπάρχουσα κατάσταση. Τώρα θέσατε το ερώτημα. Ξέρετε, είναι δύσκολο να ανταγωνιστούμε τις μπανάνες ε, των χωρών της Νίκης Αμερικής με βάση τα μέσα που έχουν τις επιφάνειες καλλιέργειας και δεν έχει καμία σχέση γενικά το προϊόν, διότι σε εμά η μπανάνα. Εμείς έχουμε περίπου ένα εκατομμύριο τόνους. Αυτοί έχουν 5-6 εκατομμύρια. Μια μικρή Λοιπόν, διακύμαση στην τιμή έχει τεράστιες επιπτώσεις. Το να πούμε λοιπόν ότι θα βρούμε ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ των δύο είναι δύσκολο. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να παραμείνει αυτός ο κλάδος βιώσιμος. Και όπως είπε η πρόεδρος, σε χώρες όπως η δική μου, όπως το Καμερούν, την μπανάνα την καλλιεργούμε σε περιοχές της υπαίθρου ε, στην οποία συμμετέχουν στην καλλιέργεια αυτή πολλοί εργάτες, μεγάλο εργατικό δυναμικό που δεν έχει άλλες δεξιότητες. Παίζει ένα πολύ έντονο κοινωνικό ρόλο αυτός ο κλάδος. Εγώ στο Τζουμπέ, στο Καμερούν επισκέφθηκα ε, μια τέτοια κοινότητα όπου υπάρχουν και σχολεία, υπάρχουν και νοσοκομεία τα οποία τα χρηματοδοτούν μέσω αυτής της δραστηριότητας. Είναι λοιπόν κρίσιμος αυτός ο κλάδος για την εργασία, για τα έσοδα, και μπορούν έτσι να συνεργαστούν πολλοί εργαζόμενοι ακόμα και με μικρό επίπεδο δεξιοτήτων. Γι' αυτό επιμένουμε. Τώρα για το Brexit. Είναι αλήθεια ότι πριν από δύο εβδομάδες είχαμε μια συζήτηση σε επίπεδο χωρώνα και ήρθε ένας εμπειρογνώμονας, ε, ο κ. Γκάρισον, ο οποίος μας εξήγησε ε, τον ε, ε, υποδεχθήκαμε, μας είπε για την Καραϊβική, μας είπε για την αγορά. 17% της δικής μας παραγωγής και της δικής μας του Καμερούν εξάγεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι. Προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε διμερές επίπεδο το Καμερούν ε, συνάντησε τις Βρετανικές αρχές που μας πρότειναν να υπογράψουμε κάποιες συμφωνίες και στο πέδο ΑΚΕ ήρθε ο Γενικός Γραμματέας του Commonwealth καθώς και ο πρέσβης που μας είπε ότι τα όποια πλεονεκτήματα ισχύουν αυτή τη στιγμή στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουν να ισχύουν. Βεβαίω, ε, είμαστε όλοι στην αναμονή αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε για την ώρα. Ξέρω ότι κάποιε χώρε πάντω, όπω και η δική μου, έχουν ξεκινήσει συζητήσει σε εμπορικό επίπεδο με το Μένο Βασίλειο για το τι θα συμβεί μετά τον Brexit σε ό,τι φορά τι εμπορικέ μα σχέσει. Αυτά μπορώ να σας απαντήσω. Οι χώρε καραβικής Καραβική βεβαίω αυτέ που επηρεάζονται περισσότερο και όχι μόνο για την μπανάνα, για πολλά άλλα προϊόντα όπου το Μένο Βασίλειο είναι η βασική αγορά για αυτούς. Ελπίζω να απάντησα στα ερωτήματά σας. Ναι βεβαίως απαντήσατε σαφέστατα κύριε Πρέσβη στα ερωτήματα που σας τέθηκαν να πω ότι βεβαίω προεδρεύω αυτή τη επιτροπή, αλλά προεδρεύω και μια μικρή ομάδα εργασία για το δίκαιο εμπόριο. Έγινε και ένα δεκαπενθήμερο την, την, ε, αυτό το διάστημα στο Μένο Βασίλειο και βεβαίω η μπανάνα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά το δίκαιο εμπόριο. Ε, κάποια σούπερ μάρκετ αγοράζουν μόνο μπανάνες από δίκαιο εμπόριο στην προέλευση στην Καραϊβική. Το θέμα του Brexit εδώ παίζει ρόλο. Ε, το θέμα της πρόσβασης στην αγορά, δηλαδή παίζει ρόλο και για το δίκαιο εμπόριο. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Να σας πω κύριε Πρέσβη, ότι η βασική μου απάντηση, μας ζητήσατε, μας λέτε, ότι δεν ζητάτε νέα γενιά συνοδευτικών μέτρων. Ε, Θέλετε απλώ η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να έχει το θέμα της μπανάνας στην μέσα διάταξη. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των δασμών. Ε, ορισμένα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Η δέσμευση τη Κομισιόν, παραδείγματο χάρη. Όποιο λοιπόν και αν προεδρεύσει τη Επιτροπή μα μετά το καλοκαίρι, μετά τι ευρωεκλογέ, ε, φαντάζομαι θα συνεχίσει να εξετάζει το θέμα τη μπανάνα, να παραμένει δηλαδή το θέμα αυτό στη μέση διάταξη, διότι με τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση η δημιουργία θέσεων απασχόληση, η δημιουργία ε, και η στήριξη τομέων που ε, βοηθούν στην ανάπτυξη του Καμερούν και άλλων χωρών τη Αφρική. Σα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ μαζί μα σήμερα. Για να ευχαριστήσω βεβαίω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι απαντήσει αλλά και για τα μέλη του Αφρό Μπανάν που είναι εδώ μαζί μας και που μας έχουν βοηθήσει και στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή και ελπίζω να έχω την ευκαιρία να έρθω να σας παρουσιάσω την άποψή μου και στο μέλλον για μια σειρά από σημεία. όπω είπα, εσεί το συνοψίσατε ήδη πολύ καλά, συνοψίσατε πολύ καλά τι ε, προσδοκίε μα μας. Θέλουμε η μπανάνα να μείνει στην ατζέντα, δεν θέλουμε δεύτερο πακέτο μέτρων, θέλουμε όμω να παραμείνει υποστήριξη, η στήριξη του τομέα και να παραμείνει αυτά τα 70 ευρώ τόνο. Ε, αν πάμε κάτω από αυτό το κατόφλι, τελείωσε ο κλάδος. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Okay, colleagues, we'll move on to items. Συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Πάμε στο σημείο 7. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Πολύ σημαντικό σημείο. Γιατί ούτως ή άλλως στην Επιτροπή μας δουλεύουμε για την αναπτυξιακή πολιτική, οπότε καλό θα είναι να μην ε, υπονομεύουμε ε, τις πολιτικές μας οι διάφορες επιτροπές. Θέλουμε οριζόντιες πολιτικές έτσι ώστε να υπάρχει συνοχή στην αναπτυξιακή πολιτική και σε όλες τις ε, διαστάσεις που την αποτελούν. Έχουμε λοιπόν την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία υποβάλλεται κάθε δύο χρόνια. Η τελευταία ήταν τον Αύγουστο του 2015. Και επειδή έχουμε αυτό το κενό, είναι επειδή η Κομισιόν ε, κινείται περισσότερο προς τους ε, ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και βεβαίως θα πρέπει αυτοί να αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της αναπτυξιακής πολιτικής γιατί οι στόχοι αυτοί αποτελούν στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. Οπότε θα κάνουμε σήμερα τη συζήτηση για το κείμενο αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την βιώσιμη Ευρώπη μέχρι το 2030 και θα ψηφίσουμε αύριο το πρωί στις 9 στην σχετική έκθεση, την σχετική έκθεση για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. έγινε μια αξιολόγηση το, της έκθεσης αυτής του 2016 που λέει ότι πρέπει να υπάρχει νέα προσέγγιση για την ε, ε, συνοχή της αναδεξιακής πολιτικής, οπότε χωρίς άλλη καθυστέρηση να δώσω το λόγο στον κύριο Μαστροτζάκομο, αναπληρωτή διευθυντή Τη ε, μονάδα για την Αναπτυξιακή Πολιτική στη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ. Σα δίνω το λόγο για να μα παρουσιάσετε την προσέγγιση τη ε, Κομισιόν και χαίρομαι που είναι εδώ και ο εισηγητή μα. Είναι εισηγητή από το 2014 και ασχολείται με τα θέματα συνοχή τη αναπτυξιακή πολιτική. Αλλά πρώτα να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μα εξηγήσει το σκεπτικό τη, τι γίνεται, που είμαστε και πώ σκέφτονται να το προχωρήσουν στο μέλλον. Σα ακούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας ε, καλέσατε να παρουσιάσουμε την έκθεση αυτή, συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής. είναι η, την έκθεση PCD. Είναι η πρώτη μετά από αρκετά χρόνια και ο λόγος για τον οποίο έχει υπάρξει αυτό το κενό στην υποβολή των εκθέσεων για τον BCD είναι ότι με την ε, υιοθέτηση της ατζέντα για το, το θεματολογίο του 2030 και την αναπτυξιακή πολιτική και τα όσα συνέβησαν το 2017, ε, πρέπει να αναθεωρήσουμε την προσέγγισή μας για τον BCD Και να εξασφαλίσουμε ότι η ε, συνοχή στην αναπτυξιακή πολιτική θα αποτελέσει την διεπαφή μεταξύ της αναπτυξιακής πολιτικής και των εσωτερικών πολιτικών. Υπάρχει ανάγκη να εξασφαλίσουμε το σχετικό άρθρο, την εφαρμογή μάλλον, του σχετικού άρθρου τη ε, συνθήκης ε, που μα ζητά να λαμβάνουμε υπόψη τον αντίκτυπο όλων των πολιτικών στις ευρωπαϊκές χώρες και για να γίνει αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το νέο θεματολόγιο που έχουμε, το περίπλοκο και το οποίο θέλουμε όλοι να υποστηρίξουμε. Και γι' αυτό έχουμε αυτή τη νέα έκθεση BCD, η οποία συνδέεται πάρα πολύ με το ε, έγγραφο στοχασμού, το οποίο υιοθετήθηκε ταυτόχρονα σχεδόν με την έκθεση BCD και το οποίο στόχο έχει να μελετήσει το πώς ακριβώς θα εφαρμόσουμε το θεματολόγιο συνολικά. Και μελετά και αυτή την, αυτόν τον ενδιάμεσο ρόλο που θα παίξει η συνοχή. Και βεβαίως η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής μπορεί να παίξει σημαντικά, σημαντικό ρόλο. Τώρα, για τούτη την έκθεση συγκεκριμένα, θα παρουσιάσω πολύ σύντομα τους βασικούς στόχους αυτής της έκθεσης, την δομή, το περιεχόμενό της και θα κλείσω με κάποια λόγια για το ποια είναι τα ευρήματα. Λοιπόν, για τους στόχους. Είναι μια έκθεση, άρα ο πρώτος στόχος είναι να κάνει έναν απολογισμό του τι έχουμε κάνει για την εφαρμογή των δεσμεύσεων BCD τα τελευταία τρία χρόνια από το 2015 όπου δημοσιεύθηκε η τελευταία μας έκθεση. Δεύτερος στόχος είναι να λάβουμε πλήρως υπόψη τις αλλαγές που έχουν υπάρξει σε παγκόσμιο επίπεδο με την υιοθέτηση του θεματολογίου και να εξάγουμε και κάποια συμπεράσματα. σχετικά με το συγκεκριμένο αντίκτυπο των αλλαγών αυτών στη δουλειά μας. Και τρίτον, να προσαρμόσουμε την προσέγγισή μας και να διευρύνουμε την έκθεση αυτή σε όλους τους ε, τομείς που ε, εμπίπτουν στην, ε, στο θεματολόγιο 2030. Είχαμε ένα μηχανισμό υποβολής εκθέσεων για, για πέντε συγκεκριμένα προεπιλεγμένα θέματα. Τώρα προσπαθούμε να μετακινηθούμε προς ένα νέο σύστημα που θα λαμβάνει υπόψη όλο το θεματολόγιο. Αυτή είναι η βασική στόχη λοιπόν Τη έκθεση. Τώρα, για τη δομή και το περιεχόμενό της. Καταρχά, υπάρχει ένα πρώτο κεφάλαιο όπου βλέπουμε αυτόν ακριβώς το σύνδεσμο της ε, συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής με τη συνολική εφαρμογή του θεματολογίου. Και γι' αυτό εξηγούμε και το ευρύτερο πλαίσιο και τη δουλειά δηλαδή που έγινε και που μας οδήγησε τελικά στο υιοθέτηση του κειμένου στοχασμού, και που μετά από κάποιες επαφές για κάποια χρόνια με διάφορες πλατφόρμες, εμπλεκόμενους φορείς λοιπά, Είχαμε και την εξωτερική αξιολόγηση που είπατε κυρία Πρόεδρε και εσείς και μας οδήγησε στη νέα έκθεση για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε δηλαδή αυτή τη νέα προσέγγιση και τον νέο αυτό τρόπο εφαρμογής. Δεύτερο κεφάλαιο που έχει μπει υπό το κεφάλαιο εταιρική σχέση, σύμπραξη, μελετά το πώς θα αλλάξουμε μηχανισμούς και εργαλεία για να εφαρμόσουμε την αυτή προσέγγιση για το BCD. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε δημιουργήσει ομάδες επιτρόπων που δουλεύουν υπό την ηγεσία του Αντιπρόεδρου Τίμερ για να δούνε τις, ε, τον αντίκτυπο της, ε, του θεματολογίου για το 2030. Επίσης, σε επίπεδο υπηρεσιών έχουμε μια διεπηρεσιακή ομάδα που ασχολείται με τους ε, στόχους της αναπτυξιακής ανάπτυξη στόχους της ανάπτυξης, βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι τακτική η παρουσία τη διπηρεσιακή αυτή ομάδα στι συναντήσει. Έχουμε επίση τροποποιήσει τα μέσα που έχουμε για την καλύτερη διακυβέρνηση. Έχουμε υιοθετήσει κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ ήδη από το 2015 και πιο πρόσφατα επίση το 2017 τροποποιήσαμε τι κατευθυντήριε αυτέ γραμμέ για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι το BCD θα λαμβάνεται πλήρως υπόψη. Έχουμε αυξήσει την ε, διάδραση με τις ε, αντιπροσωπείες, έχουν πιο ενεργό ρόλο χρησιμοποιούμε τους εξωτερικούς, ε, τους, ε, τις εκθέσεις αξιολόγηση από τις εξωτερικές υπηρεσίες για να έχουμε feedback για το τι γίνεται. Έχουμε κάνει διάφορες δραστηριότητε μέσω του BCD ε, και των σημείων επαφής για να είμαστε πιο κοντά στα κράτη-μέλη. Βεβαίως υπάρχει και η δραστηριότητα του Κοινοβουλίου στο αντίστοιχο επίπεδο τον, υπάρχει ο διορισμό ενό μόνιμου εισηγητού που μα χαροποίησε πολύ. Το BCD αναφέρεται σε διάφορα ψηφίσματα. Υπάρχουν κοινέ συναντήσει επιτροπών. Το ίδιο και στο Συμβούλιο έχει υπάρξει η ε, ομάδα εργασία που ασχολείται με την εφαρμογή της, ε, του θεματολογίου και επίση πολλά κράτη-μέλη έχουν συμμετάσχει στην ε, εκπόνηση αυτή τη έκθεση μέσω του ερωτηματολογίου που του στείλαμε πέρσι και που έτσι μπορέσαμε να λάβουμε υπόψη και την εμπειρία των κρατών μελών. Μετά, κεφάλαιο 3. Βλέπουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες BCD. Βλέπετε ότι ε, ξεπερνούμε τους πέντε παραδοσιακούς τομείς, BCD, συνοχής, αναπτυξιακής πολιτικής, και περνούμε σε μια σειρά στοιχείων που μπορεί να είναι σχετικά με τον BCD. Ας πούμε, ε, μεταρρύθμιση της κοινή ευρωτικής πολιτικής, το θεματολόγιο για τη μετανάστευση, το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Εξηγούμε τι κάνουμε σε όλους αυτούς τους τομείς και στο εμπόριο βεβαίως, χρησιμοποιώντας τα μέσα που μας δίνει το θεματολόγιο το 2030 για να δείξουμε ότι το BCD είναι ένας από τους πιο βασικούς τρόπους για να εφαρμοστεί πλήρως το θεματολόγιο. Αυτά για τη δομή και για το περιεχόμενο. Τα βασικά ευρήματα τώρα της έκθεσης. Η έκθεση αυτή δείχνει καταρχάς ξεκάθαρα ότι η πολιτική βούληση είναι κρίσιμη σημασία για να εφαρμοστεί το BCD. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για όλους μας να λάβουμε υπόψη τον αντίκτυπο των πολιτικών που χαράσουμε για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και αυτό σχετίζεται και με ένα δεύτερο βασικό έβριμα που θέλω να αναφέρω και που είναι το ότι στο νέο πλαίσιο η συνοχή για την αναπτυξιακή πολιτική σημαίνει κάτι διαφορετικό πια, κάτι καινούριο, γιατί σχετίζεται με, την, ε, αυτό που το θεματολόγιο του 2030 αναφέρει την ε, ε, συνοχή για την αναπτυξιακή πολιτική. Εμείς θέλουμε να για τους ε, στόχους της χιλιετίας, συγγνώμη. Ε, Εμεί θέλουμε να συνεχίσουμε βεβαίω να λαμβάνουμε υπόψη τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών στι πολιτικέ μα, αλλά το νέο θεματολόγιο 2030 μα ζητά να λάβουμε πιο ευρεία θεώρηση των πολιτικών που, μπορεί, που μπορούν όντω να έχουν ε, παγκόσμιο αντίκτυπο στην, στην βιώσιμη ανάπτυξη, οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά. Οπότε έτσι δίνουμε μια νέα έννοια στο BCD. Και τέλος, το τρίτο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι η σύνδεση που υπάρχει με τις τρέχουσες συζητήσεις για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, έτσι ώστε όλα αυτά να είναι συγκεκριμένα και απτά. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα μας τα ε, μέτρα, τα οικονομικά, τα χρηματοπιστωτικά θα είναι συμβατά με τον BCD, έτσι ώστε το BCD να μην θεωρείται απλώ αναπτυξιακό όργανο, αλλά να μπορεί να συμβάλλει στην χάραξη πολιτική συνολικά. Και, αυτός βεβαίως, ε, και αυτό το σημείο είναι ένα σημείο στο οποίο ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σημαντικό. Τέλο, κυρία Πρόεδρε, να πω δύο πράγματα για την εξωτερική αξιολόγηση του BCD που συνδέεται στενά, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια εξωτερική αξιολόγηση για την εφαρμογή της πολιτικής BCD από το 2009 μέχρι το 2016. Έχει γίνει λοιπόν αυτή η εξωτερική αξιολόγηση, πρόσφατα δημοσιεύθηκε και τώρα θα δώσουμε και εμείς τη δική μας άποψη μέσω ενός staff working document, το οποίο θα υιοθετηθεί σύντομα, όπου θα δούμε ποια είναι τα ευρήματα και οι συστάσεις της αξιολόγησης και θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πώς έχουμε έστω και μερικώς εφαρμόσει ε, κάποια από αυτά που ζητά να γίνουν η ε, εξωτερική αξιολόγηση. Και πώς επίσης ε, θα φροντίσουμε να ακολουθήσουμε τις συστάσεις τους. Νομίζω ότι μπορώ να σταματήσω εδώ. Πρόεδρε, αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ έχω μια-δυο ερωτήσεις, αλλά καταρχάς θα δώσω το λόγο στον κύριο Πρέντα, που είναι ο μόνιμος μας ε, εισηγητής. Ευχαριστώ, Λίντα. Ναι, ε, είμαι μέσα στον ήλιο. Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Νόιζερ που είναι εδώ σήμερα για να συζητήσουμε το ΠΣΔ. πρόκειται για έναν ε, σημαντικό θεσμό που όμως λειτουργεί ε, Λειτουργούμε μάλλον συγγνώμη στο μίνιμουμ. Ε, ε, μόνο δύο είμαστε παρόντες. Δείχνει αυτό και το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε άλλωστε. Είμαι ικανοποιημένο που ήρθατε, γιατί περιμέναμε πολύ καιρό. Καταλάβαμε ποια ήταν η στρατηγική. Βεβαίως ε, καταλαβαίνουμε ποια είναι η στρατηγική. Εν ώψη του εκλογικού χρονοδιαγράμματος ε, φέτος δεν μπορούμε να απαντήσουμε επισήμως σε αυτή την έκθεση. Αυτή η τελεγή απόψεων είναι μια ευκαιρία για να κάνουμε έναν απολογισμό για την ε, συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών. Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2015. Εντάξει, φτάνει μέχρι εκεί που κατεβάσατε τα σκέστα. Δεν χρειάζεται να κλείσουμε και όλη την, μέρα, την όμορφη αυτή μέρα έξω. Εντάξει, Κριστιαν, μπορείς να συνεχίσεις. Βεβαίω περιμέναμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή μια νέα έκθεση, διότι θέλαμε επισήμως να καταστούν σαφή τα πράγματα, δηλαδή και οι δύο πολιτικές για την συνοχή των, πολιτικών, των αναπτυξιακών πολιτικών και την συνοχή για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ακόμα και αν είχαμε τη συνένεση ε, που μιλήσαμε ήδη για το 2000, μέχρι το 2030. Εκτιμώ το γεγονός ότι η συνοχή των απταξικών πολιτικών αποτελεί νομική υποχρέωση και προτεραιότητα και ακόμα και αν τα κράτη-μέλη μας έχουν ακόμα πολλά να κάνουν όσον αφορά την εναρμόνιση των πρακτικών τους. Η έκθεσή σας αποκαλύπτει ότι ορισμένοι αντικατέστησαν την PCD από την PCSD και ελπίζω πως αυτό δεν θα αποδυναμώσει την έννοια του αυτής της υπόθεσης ε, Υπήρξαν πρόοδοι βεβαίω και θέλω να αναφέρω δύο συγκεκριμένα σημεία που θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι η πιο συστηματική χρήση των αναλύσεων αντικτύπου στην ε, σύλληψη των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ληφθούν υπόψη να ληφθεί υπόψη οι πιθανές συνέπειες για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεύτερο θετικό στοιχείο, δεύτερη πρόοδος είναι η ε, πιο σημαντική συμμετοχή των ε, εμπλοκή των ευρωπαϊκών αντιπροσωπιών. Η ανταλλαγή επιρρεών και ο διάλογος που θέσπισαν με τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι μέσα απαραίτητα για να προχωρήσει η ε, συνοχή αυτή. Και μάλιστα με χαρά διαπίστωσα ότι έχει δημοσιευθεί και μια εξωτερική αξιολόγηση της ε, PCD. Το είχαμε ζητήσει αυτό και παλιότερα. Ε, Λυπούμε λοιπόν, ωστόσο που τα στοιχεία που αφορούν την περίοδο 2009 2016 δημοσιεύθηκαν μόλις φέτος. Δηλαδή μιλάμε φέτος για το τι συνέβη πριν 10 χρόνια. Κάλλιο αργά παρά ποτέ λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάπω αργά. Ε, η, η πολιτική αυτή είναι περίπλοκη έννοια και δεν διευκολύνει πραγματικά τα πράγματα. Ε, βρίσκουμε εδώ στοιχεία τα οποία εγώ είχα συμπεριλάβει στην έκθεσή μου το 2016. Το θέμα του modus operandi, του μηχανισμού της ε, PSD, το τι κάνει ποιος μέσα στους θεσμούς. Είναι προφανές πως η Κομισιόν δεν πρέπει να δίνει οδηγίες στις άλλους θεσμούς σε σχέση με την ε, PSD, αλλά μπορεί να δώσει σαφείς προσανατολισμούς. Δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο αξιολόγησης είναι πώς τα μέσα της PSD θα επηρεάσουν άμεσα τη... τις πολιτικές. Μα ποιος παίζει με τα σκίαστρα, διακόπτει ο κ. Όλοι γνωρίζουμε ότι ε, πρέπει να βρούμε τρόπο να προχωρήσει αυτή η PSD και ελπίζω πως η απάντηση της Κομισιόν θα μπορέσει να μας δώσει λαβές για ενδιαφέροντα προβληματισμό και για τα επόμενα χρόνια, γιατί αν η εφαρμογή των στόχων και μέχρι το 2030 είναι μεν προτεραιότητα, η δεν πρέπει να βρει τη θέση της και να αξιοποιήσει τα ατού της για να συμβάλλει στην λειτουργική χρήση της PSSD. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όσους θα είναι στην επόμενη θητεία στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Τα έχουν περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Και ζητώ συγγνώμη για το πρόβλημα με τα σκίαστρα. Από ό,τι κατάλαβα πάνε πάνω ή κάτω, δεν μπορούν να σταματήσουν στη μέση. Αυτό είναι το θέμα. Συμφωνώ μαζί σας που είμαστε τόσο λίγοι σήμερα εδώ. Είναι λυπηρό, αλλά επειδή έρχονται εκλογέ. Αυτοί που δεν έρχονται, δεν επιστρέφουν, ε, ασχολούνται με άλλα θέματα και αυτοί που θέλουν να επιστρέψουν ασχολούνται ήδη με την εκστρατεία. ναι, μόνο κάποιες παρατηρήσεις έχω να κάνω. Ευχαριστώ τον Σκιώδη Έχουμε και την μήνυ σύνοδο, γι' αυτό είναι έτσι τα πράγματα. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε μία πιο ε, σταθερή συζήτηση, γιατί έχει φτιαχτεί η PCD, αλλά το μέγα πρόβλημα κατά τη γνώμη μου είναι πώς θα μπορέσουμε καλύτερα να επηρεάσουμε όσον αφορά τη λήψη πραγματικών αποφάσεων στις άλλες επιτροπές. Ε, επειδή ακριβώς όμως εμείς είμαστε εδώ παρόντες, δραστήριοι, ε, ίσως και να επανεκλεγούμε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ Νόρμπετ. Εγώ θέλω να ρωτήσω μια ερώτηση την Κομισιόν, ίσως να μην αφορά όμως μόνο την DGFCO. Όταν ε, συνομιλώ με το κοινό μιλούν για την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική που, και για πράγματα που αλήθευαν πριν από λίγα χρόνια, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ τα τελευταία 15 χρόνια. Ήταν προβλήματα παλιότερα, αλλά τώρα έχουν λυθεί λόγω των προσπαθειών που έχουν γίνει. Ένα παράδειγμα είναι η κοινή αλληλευτική πολιτική, η οποία έχει βελτιωθεί πολύ όσον αφορά τι αναπτυξιακέ πτυχέ. Δεν είναι τέλεια, αλλά έχει βελτιωθεί πολύ. Διερωτώ με λοιπόν, εντάξει, αυτά τα έγγραφα είναι μακροσκελή, δι, ε, ε, δεν είναι γλώσσα δηλαδή που ο κόσμος καταλαβαίνει εύκολα. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να κάνει κανείς όπως και ο Νόρμπερ, γιατί σε άλλες επιτροπές στη Not Financial Reporting υπάρχουν βήματα που έχουν γίνει όσον, όσον αφορά τη διαφάνεια. Εν πάση περιπτώσει, ξέρω ότι και αυτή εδώ η έκθεση είναι πολύ μακροσκελή και δεν είναι, σαφής, δεν είναι σαφές ποια είναι τα μεγάλα επιτεύγματα της Κομισιόν όσον αφορά την PCT και ποια είναι οι μεγάλες προκλήσεις που μας περιμένουν, πού υπάρχουν τα κενά. Εγώ θα ήθελα κάπου να μπορώ να δω σύντομα τι ακριβώς ε, ισχύει και συμβαίνει. Να έχουμε μια αξιολόγηση, εκεί που τα πήγαμε καλά να το λέμε δηλαδή. και να συγκρίνουμε και με άλλα μέρη του κόσμου. Να είμαστε περήφανοι για το τι έχουμε κάνει, αλλά και σαφείς για το τι ακόμα πρέπει να γίνει. Γιατί πολλές φορές σε αυτές τις εκθέσεις έχουμε τόσο πολλές λεπτομέρειες που το ουσιαστικό μήνυμα χάνεται. Και ε, όπως είπα, να, αυτό να φαίνεται κάπως καλύτερα, πού έχουμε προοδεύσει και πού πρέπει να τα πάμε καλύτερα. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ακούστε, το πρώτο που ήθελα να πω είναι αυτό που είπε και ο εισηγητής για το PCD και το PCSD. Είναι αυτό που σκεφτόμαστε ακριβώς και εμείς. Δηλαδή, βεβαίως και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τη νέα ατζέντα και το πόσο περίπλοκα είναι τα ζητήματα αυτά. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε τον στόχο του άρθρου 208 και την ιδιαιτερότητα της πολιτικής αυτής ε, της αναπτυξιακής βοήθειας. Ε, και μας λοιπόν μας απογοήτευσε κάπως το γεγονός ότι κάποια κράτη-μέλη από ό,τι φαίνεται θεωρούν ότι στο νέο πλαίσιο μπορούμε να ξεχάσουμε την PCD και μπορούμε να εργαστούμε πάνω σε μια ευρύτερη έννοια που δεν εξετάζει απαραίτητα τα συμφέροντα ε, των αναπτυσσόμενων χωρών. Εμεί πιστεύουμε ότι εξακολουθεί να είναι κρίσιμο να συμβεί κάτι τέτοιο και προς την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Γι' αυτό που το, το, το χρονοδιάγραμμα που κ. Μπρέντα είναι σημαντικό Βεβαίω. Υπάρχει όμω και κάτι θετικό εδώ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια καλή συγκυρία. Δημοσιεύουμε αυτό το έγγραφο, σύντομα δημοσιεύουμε ένα άλλο για την αξιολόγηση. Είναι ακριβώς η στιγμή που θα συζητήσει το Συμβούλιο, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το έγγραφο διαβούλευση. Θα είμαστε λοιπόν έτσι σε θέση να πιέσουμε κάπω για τα δικά μα θέματα τη PCD είναι αυτή τη στιγμή επίκαιρα αν θέλετε. Γι' αυτό που είπατε τώρα για την επικοινωνία κυρία Πρόεδρε, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι και αυτό βέβαια περίπλοκο ζήτημα ε, σε σχέση με τον αντίκτυπο δηλαδή των εργασιών μας σε μια σειρά τομείς. Είχαμε αρχίσει να δουλεύουμε πάνω σε ένα σχέδιο επικοινωνιακό. Θελήσαμε να ετοιμάσουμε ε, κάποιο φυλάδιο με κάποια γραφήματα που να είναι φιλικό, φιλικά προς το χρήστη και που τα εξηγούν με λίγα λόγια ε, ποιες, ε, ποιοι είναι οι βασικοί τομείς όπου θεωρούμε ότι ελήφθη με επιτυχία υπόψη η πολιτική συνοχής για την ανάπτυξη ελπίζω να μπορέσουμε να σας δείξουμε τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών σύντομα. Τώρα για τις μελλοντικέ προκλήσεις. Βεβαίω είναι πάντα δύσκολο αυτό το ερώτημα. Αυτό που έχει σημασία πιστεύω είναι να αντιληφθούμε ότι η δουλειά γύρω από το θέμα της συνοχής της πολιτικής ε, είναι μια δουλειά η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Ε, πάντα θα προκύπτουν θέματα όπου θα πρέπει να εξετάζουμε το, τον ενδεχόμενο αντίκτυπο ε, και να αξιολογούμε αυτόν τον αντίκτυπο σε διάφορους ε, ε, σε διάφορους τομείς που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, την βιώσιμη ανάπτυξη, την αναπτυξιακή βοήθεια. Η πρόκληση λοιπόν είναι να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε μόνιμη βάση. Και όπως είπε και ο εισηγητής, η νέα μορφή ε, του αντικτύπου μας βοηθάει για να το κάνουμε αυτό και η δουλειά που κάνουμε ε, στην Κομισιόν στα πλαίσια της ατζέντας για το 2020-2030 ε, μπορούμε έτσι με οριζόντιο τρόπο ε, να εμπλέξουμε όλες τις κοινικές διευθύνσεις ε, που παίζουν ρόλο στα ζητήματα αυτά. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Καλώς, καλώς ήρθατε κυρία Σόνικ. Ε, λοιπόν, δεν βλέπω να θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Ναι, θα ήθελα, ε, είναι σίγουρα η τελευταία φορά που θα συζητήσουμε την πολιτική, συνοχή της πολιτικής την ανάπτυξη, ε, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πρέντα πάνω απ' όλα από το 2014 για τη δουλειά του εδώ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερο, μεγαλύτερη συμμετοχή για την τελευταία συνάντηση, αλλά είναι εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι εδώ και στην επόμενη θητεία και είναι αυτοί που μετράνε. Να ευχαριστήσουμε τον Κρίστιαν και να το χειροκροτήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Συνάδελφοι, τώρα ολοκληρώνουν οι εργασίε μας για σήμερα. Τώρα είναι το θέμα των συντονιστών. Θα μπορούσαμε να αρχίσουμε μέσω με του συντονιστέ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται αυτό. Οπότε 5 και μισή. Ε, στείλτε πάντως τα μηνύματα στους συντονιστές. Ε, εγώ θα, είμαι, θα ξεκινήσω 5 και μισή ακριβώς. Δεν έχουμε και πολλά να συζητήσουμε και σε 20 λεπτά θα έχουμε τελειώσει. Είναι ένα όμορφο απόγευμα και αύριο θα αλλάξει ο καιρός. Οπότε καλό είναι να μπορέσετε σήμερα να αποφεληθείτε. 5.30 ακριβώς θα αρχίσουμε λοιπόν. 9 η ώρα αύριο ψηφίζουμε. Α, βλέπω ότι αλλά άλλαξε πάλι. Στο 2Q2 γίνεται από κοινού με την Επιτροπή ΕΜΒΗ η ψηφοφορία. 2Q2 καλό είναι να στείλουμε κάποιο μήνυμα διότι υπήρξε σύγχυση σήμερα ε, ότι ξεκινάμε 9 στο 2Q2 έτσι διότι σήμερα το απόγευμα και εγώ μπερδεύτηκα, χάθηκα, συνάντησα τον Νόρμπερτ. Ε, να θυμίσουμε λοιπόν 2Q2 και μετά εδώ για συζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους, θα τα πούμε αύριο με τους υπόλοιπους. Γεια σας.